θα θεωρηθούν εγκεκριμένοι και αυτοί οι διορισμοί. Δύο γραπτές αιτήσει ε, υποβλήθηκαν και υπογράφηκαν από δύο μέλη του Κοινοβουλίου της κυρία Ελένα Τζεντήλ και άλλων 15 μελών για τις ιδιοπαθή ε, ανακοίνωση και ο κύριος ε, Λουί Μισελ και άλλα 11 μέλη υπέγραψαν ε, έτοιμα για την αφαίρεση οργάνων ε, στην Κίνα. Οι δηλώσεις αυτές θα δημοσιευτούν μαζί με τα ονόματα των όσων προσυπέγραψαν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Erklärung zur